Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, έχουμε τι προφορικέ ερωτήσει προ την Επιτροπή ε, και το Συμβούλιο για την εξάλληψη τη βία εναντίον των γυναικών. Σα υπενθυμίζω ότι σήμερα είναι η διεθνή ημέρα για την εξάλληψη τη βία εναντίον των γυναικών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η συζήτηση για μα αποτελεί μια πολύ σημαντική ευκαιρία. Δίνω λοιπόν ευθύ εξ αρχή ε, το λόγο στην κυρία Σβένσον, την εισηγήτρια, για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι σήμερα είναι 25η Νοεμβρίου, η δεκάτη επέτειος της Παγκόσμιας ημέρας του ΟΗΕ για την βία κατά των γυναικών για την καταπολέμηση μάλλον αυτή της βίας. Σε όλη μου την ενήλικη ζωή πρέπει να σας πω ότι έχω εργαστεί σε γυναικείες οργανώσεις και σε δίκτυα για την καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών. Πιστεύω λοιπόν ότι στη διαδρομή της εργασίας μου μπόρεσα να χρησιμοποιήσω σαφή ορολογία για να διατυπώσω πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Λόγια, λόγια, λόγια. Επανειλημμένα λέμε τα ίδια πράγματα. Και πραγματικά ήρθε η ώρα για απτά μέτρα. Διότι η βία στερεί, κλέβει τα ανθρώπινα δικαιώματα από τις γυναίκες. Επηρεάζει την καθημερινότητά τους και η βία σίγουρα προσδιορίζει την ζωή των νέων γυναικών. Όλοι έχουμε λοιπόν ευθύνη για να σταματήσει αυτή η εκοφαντική σιωπή. Πρέπει να συνεργαστούμε και εντός και εκτός της κοινοβουλευτικής συνέλευσης με όλες τις δυνάμεις για να σπάσουμε τον κύκλο της βίας. Της βίας είτε είναι σεξουαλική, είτε είναι ψυχολογική, είτε πρόκειται για βιασμούς, είτε πρόκειται για δουλεία, για πορνεία, ε, για ακροτισμούς των γεννητικών αργάνων. Είναι ένα όπλο ακόμη και στις συγκρούσεις και στους πολέμους. Πρέπει να ενεργήσουμε συλλογικά και ατομικά κατά της βίας. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι η βία στις οικογενειακές σχέσεις είναι ιδιωτική υπόθεση. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Ε, πρόκειται για διαρθρωτική βία, είναι κοινωνικό ζήτημα. Η κοινωνία πρέπει να σταματήσει τον κύκλο της βίας όπως είπα. Είναι επεκτή εκτενές πρόβλημα σε πολλές περιοχές και σε όλες τις επίρους. Ε, πρέπει να σταματήσει κάθε μορφή βίας που έχει σχέση με το φύλλο. Αυτό είναι η θεμελιώδης αρχή της ισότητας στην κοινωνία. Η βία των ανδρών προς τις γυναίκες καταδεικνύει την ανισότητα των σχέσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ταυτόχρονα συμβάλλει στην διατήρηση των ε, σχέσεων εξουσίας που υφίστανται σήμερα. Συνεπώς, πρέπει να αγωνιστούμε για να σταματήσει η βία των ανδρών κατά των γυναικών και των κοριτσιών και η βία δεν είναι εξουσία. Μιλάμε για στερεότυπα σεξουαλικά, στερεότυπα φύλου που βασίζονται στην άποψη ότι οι άνδρες είναι ανώτεροι των γυναικών. Η βία κατά των γυναικών καταδεικνύει ακριβώς την έλλειψη ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι και θέμα δημόσιας υγείας πρέπει να πω, είναι κοινωνικό πρόβλημα. Και πέραν της προσωπικής οδύνης και του πόνου υπάρχει και ένα κόστος για την κοινωνία. Αλλά βασικά είναι θέμα ισότητας και γι' αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με αυτή την προσέγγιση. Ακόμη αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατάφερε να υιοθετήσει μέτρα. Και ακριβώς οι συνάδελφοι και εγώ ζητούμε να ληφθούν αυτά τα μέτρα. Έχουμε ήδη το πρόγραμμα Δάφνη, το οποίο δίνει κάποια οικονομική υποστήριξη σε ορισμένες πρωτοβουλίε για την καταπολέμηση της βίας. Θετικό αυτό και απαραίτητο. Αλλά παντελώς ανεπαρκές σε σχέση με τα απαιτούμενα, τα πραγματικά απαιτούμενα. Γι' αυτό η Επιτροπή των Δικαιωμάτων της των γυναικών του Ευρωκοινοβουλίου θα θέλαν να ακούσουν τι θα κάνει η Κομισιόν και το Συμβούλιο για να οδηγήσουν τα κράτη-μέλη στην δημιουργία προγραμμάτων. Υποστηρίζει η Κομισιόν τον, ένα τέτοιο σχεδιασμό, ώστε τελικά να έχουμε κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες για ένα ενιαίο στρατηγικό ευρωπαϊκό σχέδιο. Υπάρχει υποχρέωση να βοηθήσουμε την ισότητα και αυτό βρίσκεται και στις συνθήκες. Καταλήγοντας, πότε η Κομισιόν θα οργανώσει ευρωπαϊκό έτος κατά της βίας εναντίον των γυναικών. Είναι κάτι που ζητάμε συνεχώς στο Ευρωκοινοβούλιο από το 1997. Ήγκηκε η ώρα λοιπόν. Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο κύριος ε, Τόρτεν, ο κύριος Υπουργός. Η κυρία Τόρστενσον. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η πρόεδρος ε, της Επιτροπής Ισότητας και Δικαιωμάτων Γυναικών έτσι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και θέλω να ξεκαθαρίσω αμέσως πως η βία κατά των γυναικών δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Φέτος έχουμε, ρωτάζουμε την δέκατη επέτειο του ψηφίσματος του ΟΗΕ που ορίζει την 25η Νοεμβρίου ως ημέρα καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Στρέφεται σήμερα η σκέψη μας στις αμέτρητες γυναίκες που υποφέρουν στις ε, περιοχές όπου υπάρχει πόλεμος, γνωρίζουμε πως υπάρχουν γυναίκες που βιάζονται, που παρενοχλούνται, που υφίστανται βάρβαρες ε, παραδοσιακές πρακτικές. Είμαστε επίσης κατά των ε, γάμων ε, με καταναγκασμό και κατά των λεγόμενων εγκλημάτων τιμής που κυμαίνονται από ακροτηριασμό μέχρι δολοφονία. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τη βία κατά των γυναικών που διαπράττεται εις βάρος των γυναικών στην Ευρώπη σε καθημερινή βάση. Το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται σε διάφορους τομείς της πολιτικής. Αντικατοπτρίζεται αυτό ξεκάθαρα στο ψήσιμο το οποίο θα ψηφίσετε αύριο, η βία κατά των γυναικών. Δεν είναι μόνο ένα έγκλημα, και αδικία εις βάρος των γυναικών, αλλά είναι και ζήτημα των ανδρών ως εγκληματιών και ζήτημα ισότητας των ε, δύο φύλων. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση, να υπάρχει ένας ευρύτερος ορισμός ε, της βίας ε, κατά των γυναικών. Εμείς λοιπόν έχουμε καθοδηγηθεί από την αρχή της ενσωμάτωσης πολιτικής των φίλων σε όλες τις ε, πολιτικές μας. Στο άρθρο 23 της ε, συνθήκης ε, δεσμευόμαστε να προωθήσουμε την ισότητα άνδρων και γυναικών σε όλους τους τομείς πολιτικής. Το Συμβούλιο κατά καιρού έχει αναφερθεί στο πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών. Θα ήθελα να ξεκινήσω τώρα με κάτι το θετικό ένα από τα πιο επιτυχή παραδείγματα τέτοιας ενσωμάτωσης της ισότητας ήταν στο θέμα των γυναικών στις ένοπλες συγκρούσεις όπου έχουμε μια πιο συνολική πολιτική. Εξπακούεται πως ε, το Συμβούλιο περιορίζεται σε αυτά τα οποία ορίζει η συνθήκη και πως τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για τα ζητήματα που είναι δική τους αρμοδιότητα, ειδικά τα ζητήματα δικαιοσύνης και εσωτερικών και υγείας. Είναι προνόμιο των κρατών μελών να καθορίσουν τα σχέδια καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, αλλά μπορούν να εποφεληθούν από την συνεργασία και επιπλέον υπάρχουν μέτρα στο ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της βίας των και της σωματεμπορίας που είναι ένας από τους έξι τομείς που αναφέρονται κατά προτεραιότητα στον οδικό χάρτη από το 2006 έως το 2010 και σοχεύουμε να έχουμε συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία να αυξηθεί η ευαισθησία και να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές στην έρευνα. Αναμένουμε λοιπόν ένα νέο σχέδιο ισότητας για την περίοδο 2011-2015. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης που θα εγκριθεί τον επόμενο μήνα μας δίνει ένα πλαίσιο για πολλές από αυτές τις ανησυχίες που έχει εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναμένουμε κάποια συμφωνία επί του προγράμματος και επί της εφαρμογής του πολλά έχουν ήδη γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ειδικά όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών, την ευαισθητοποίηση και τις βέλτιστες πρακτικές. Κάποιοι από εσάς ήσασταν παρόντες και στο συνέδριο που έκανε η Προεδρία πρόσφατα στη Στοκχόλμη με το ίδιο θέμα. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας και να συζητήσουμε τις μελλοντικέ ε, πολιτικές. Η απόφαση του 2007 που όριζε ένα πρόγραμμα ονόματι Δάφνη 3 για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών. Είχε ζωτική σημασία. Καλωσορίζω την θετική επίδραση που είχε το πρόγραμμα Δάφνη στις ε, κοινότητές μας. Δικαίως εσείς ε, τονίσατε στο ψήφισμά σας το ότι δεν υπάρχουν συγκρίσιμα δεδομένα για τους διαφορετικούς τύπους βίας κατά των γυναικών. Το Συμβούλιο γνωρίζει πάρα πολύ καλά πως η συλλογή συγκρίσιμων και ακριβών δεδομένων είναι πολύ σημαντική για να προλάβουμε τη βία κατά των γυναικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελπίζω λοιπόν πως το μέλλον το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των δύο φίλων που έχει συσταθεί από κοινού από Κοινοβούλιο και Συμβούλιο θα συνεισφέρει σημαντικά στον ε, τομέα αυτών. Το Συμβούλιο το ίδιο έχει ήδη έχει λάβει αυτά μέτρα για να αυξηθεί η συγκρισιμότητα των δεδομένων και έχουμε εργαστεί στο πλαίσιο της πλατφόρμας του Πεκίνου και έχουμε αναπτύξει τρεις δείκτες ε, που έχουν σημασία εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα βία στο σπίτι, οικογενειακή βία, δεύτερον σεξουαλική παρνόχληση στο χώρο εργασίας και τρίτον γυναίκες στις ένοπλες συγκρούσεις. Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, αλλά προφανώς πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα. Οι πιο ευάλωτες γυναίκες ζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το γνωρίζουμε αυτό και αυτό έχουμε υιοθετήσει μια σειρά συμπερασμάτων για την ισότητα και την ενδυνάμωση των γυναικών στην αναπτυξιακή συνεργασία. Αυτό τονίζει την σημασία του να αντιμετωπίσουμε την βία εις βάρος των γυναικών και συμπεριλαμβανομένων παραδοσιακών πρακτικών όπως ο ακροτηριασμός των γενετικών οργάνων αλλά δεν θα πρέπει να μείνουμε εκεί μόνο. Ο ακροτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, τα λεγόμενα εγκλήματα τιμής, η με καταναγκασμό, είναι όλα ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν πάντα στην πρωτοπορία με το να καλεί να καταπολεμηθούν αυτές οι παραδοσιακές πρακτικές και επαναβεβαιώσαμε την δέσμευσή μας στα συμπεράσματα που υιοθετήσαμε πέρσι για, για τα κορίτσια. Και εκεί πέρα τονίζουμε και αναφέρω επιλέξει πως η εξάλληψη κάθε μορφής βίας κατά των κοριτσιών συμπεριλαμβανομένης σωματεμπορίας και λοιπόν πρακτικών είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ενδυνάμωση κοριτσιών και γυναικών και για να επιτύχουμε ισότητα ανδρών και γυναικών στην κοινωνία όπως ε, τόνισε και η κυρία Βουλευτής ε, στην εισαγωγή της ε, η βία κατά των γυναικών βλάπτει την δυνατότητά τους ε, να ασκήσουν μια ενεργή κοινωνική ζωή και οι γυναίκες οι οποίες έτσι παρεμποδίζονται από τις κοινωνικές δραστηριότητες και την δουλειά κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν και να καταλήξουν στην φτώχεια. Οπότε επανέρχομαι στην συνολική προσέγγιση για την οποία μίλησα στην αρχή. Το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών είναι ευρύτερο ε, ζήτημα ανισότητας και υπάρχει μια ευρύτερη εκστρατεία ενδυνάμωσης των γυναικών και αντιμετώπισης της βίας. Οι γυναίκες οι οποίες είναι ελεύθερες να εκδιπλώσουν το πλήρες ε, δυναμικό τους ε, είναι βεβαίως λιγότερο ευάλωτο στη βία από τις γυναίκες τις αποκλεισμένες. Επίσης η Κομισιόν τακτικά επαναλαμβάνει την ανάγκη της καταπολέμησης της στόχιας των γυναικών και βεβαίως η απασχόληση είναι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό και πρέπει να διευκολύνουμε την συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Η οικονομική και κοινωνική κρίση αυξάνει το ευάλωτο των γυναικών και βεβαίως είχαμε και τα συμπεράσματα τα σχετικά που μιλούσαν για ενίσχυση της ε, απασχόλησης των γυναικών και σχετική μνήμα στη συνθήκη της Λισαβόνας και σκοπεύουμε να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος σε ζητήματα που αφορούν τα δύο φύλλα στη μελλοντική στρατηγική. Καθώς λοιπόν εορτάζουμε την δέκατη επέτειο του ψηφίσματος του ΟΗΕ που ορίζει Διεθνή ημέρα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών αναγνωρίζουμε το εύρος του προβλήματος αλλά ταυτόχρονα καλωσορίζουμε το ότι οι χώρες συνεργάζονται για να το καταπολεμήσουν και πράγματι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας εδώ στην Ευρώπη γίνεται σε διεθνές πλαίσιο. Κατά την επόμενη συναντησή μας, το Μάρτιο του 2010, η Επιτροπή Γυναικών των Ηνωμένων Εθνών θα προβεί στην επαλήθευση, στην επαλήθευση του κατά πόσο έχει προχωρήσει το κείμενο του Πεκίνου και θα εξετάσει επίσης και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ε, προκλήσεις που πρέπει ακόμα να αντιμετωπιστούν. Στις 30 Νοεμβρίου το Συμβούλιο λοιπόν καλείται να εγκρίνει μία σειρά διατάξεων που αφορούν στο ε, πρόγραμμα του Πεκίνου. Θα μας δώσει λοιπόν μία δομή και μία μακροπρόθεσμη μερίσια διάταξη που θα αφορά στην πολιτική της ισότητας των δύο φύλων. Το Συμβούλιο λοιπόν είναι άμεσα ε, εμπλεγμένο, συμμετέχει άμεσα σε αυτή την όλη διαδικασία για να αντιμετωπιστεί η βία κατά των γυναικών. Το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών δεν περιορίζεται σε εθνικά σύνορα. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστεί σε διεθνείς φορείς τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της Ευρώπης. Οφείλουμε λοιπόν να ε, εντείνουμε τον αγώνα κατά της ε, ε, βίας εις βάρος των γυναικών και δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας μπροστά σε περιπτώσεις ε, βίας που πλήττουν τους συμπολίτες μας και που λαμβάνουν χώρα ενδεχομένω και μέσα στο σπίτι μας. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, επαναλαμβάνω αυτά που είπα στην αρχή, ότι δηλαδή η βία που ασκείται εις βάρος των γυναικών δεν μπορεί να νομιμοποιείται σε μια κοινωνία που αυτορίζεται πολιτισμένη. Είμαι ευτυχής ε, που μου δόθηκε ευκαιρία σήμερα να παρουσιάσουμε το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχετε την υποστήριξη και του Συμβουλίου και της Προεδρίας για να υπεραμεινθείτε του, ε, της αρχής ε, της ισότητας και της δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. ευχαριστούμε Υπουργέ και τώρα να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ντεκούτ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επ' ευκαιρία της ε, Παγκόσμιας ημέρας για την εξάλληψη της βίας εναντίον των γυναικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να επαναλάβει τη δέσμευσή της, την πολιτική της δέσμευση, την ισχυρότητη πολιτική της δέσμευση, ε, να αγωνιστούμε για την εξάλληψη της βίας εναντίον των γυναικών. Αυτό εκφράζεται και στην ανακοίνωση για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, που ανάμεσα στις προτεραιότητες συμπεριλαμβάνει και την ανάγκη να ε, δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα των δικαιωμάτων των παιδιών και στην προστασία των ιδιαίτερα ευάλωτων ατόμων, όπως οι γυναίκες που είναι θύματα βίας και οι ηλικιωμένοι με τον οδικό χάρτη ε, για την ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα για το χρονικό διάστημα 2006-2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να συμβάλλει στην εξάλληψη της βίας ε, που συνδέεται με το φύλλο ε, και στο εμπόριο ανθρώπων. Η καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών αποτελεί σημαντική προτεραιότητα και της νέας στρατηγικής που θα διαδεχθεί τον οδικό χάρτη και από αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας είναι εξίσου σημαντικό ε, να χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένε δράσει επιτόπου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην καταπολέμηση τη βία στην Ευρώπη διαμέσου του προγράμματο Δάφνε, Δάφνη, ε, ενώ η η απάντηση ε, σε επίπεδο πρόληψης ε, της βίας θα πρέπει να ενισχυθεί με πιο συγκεκριμένες δράσεις. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντοπίσει συγκεκριμένε δράσει στα πλαίσια του Δάφνη 3 για την υλοποίηση μια πιο συνεκτική στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση τη βία εναντίον των παιδιών, των νέων και των γυναικών. Χάρη σε ε, ετήσιο ε, προπολογισμό 17 περίπου εκατομμύρια 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στράφηκε συγκεκριμένα προ την κατεύθυνση των ομάδων που διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο και αυτό πέραν των ενισχύσεων που λαμβάνονται μέσω των εθνικών προγραμμάτων. Στα πλαίσια του προγράμματο εργασία Δάφνη 3 για το 2010, ε, σκεφτόμαστε και την δημιουργία συμβουλευτική ομάδα εμπειρογραμμόνων που θα μπορούσε να βοηθήσει για τον εντοπισμό των απαραίτητων δράσεων σε κοινοτικό επίπεδο και για την ενθάρρυνση μια κοινή προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση θα ξεκινήσει μια σημαντική μελέτη σκοπιμότητα για την αξιολόγηση του κατά πόσον θα πρέπει να, υπάρξει εναρμόνιση τη νομοθεσία κατά τη βία που, ε, με βάση ε, που, που στηρίζεται ε, λόγω φύλου μάλλον ή λόγω ηλικία και όλα αυτά θα παρουσιαστούν το φθινόπωρο 2010. Η πρόθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να συγκαλέσει του εκπροσώπου των κυβερνήσεων των κρατών μελών, των κοινοτικών θεσμών, των πολιτικών ομάδων, των οργανώσεων τη κοινωνία των πολιτών και των διεθνών οργανώσεων κλπ. με στόχο την κατάρτιση μια πιο συγκεκριμένη ε, κοινοτική πολιτική. Εξάλλου, η ανταλλαγή καλών πρακτικών ε, και ε, μοντέλων παρέμβαση ήδη αποτέλεσε αντικείμενο οργανωμένη συζήτηση το Δεκέμβριο 2007 υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Πρόληψη Εγκληματικότητα. Τέλο, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι ακραίε μορφέ βία εναντίον των γυναικών θα πρέπει να ε, καταπολεμηθούν με τα πλέον αυστηρά μέτρα. Προ την κατεύθυνση αυτή, η Επιτροπή πρότεινε το Μάρτιο τροπολογία του Ευρωπαϊκού Ποινικού Πλαισίου για την ε, τομέα καταπολέμησης του εμπορίου των ανθρώπων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών. Ε, πράγμα το οποίο αφορά ιδιαίτερα τις γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια, δηλαδή τις πιο ευάλωτες ομάδες. Όσον αφορά την, ε, ε, τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Έτους για τη βία κατά των γυναικών. Με βάση μια εις βάθος αξιολόγηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο ότι ε, θα ήταν πρόωρο ενδεχομένω να έχουμε μια τέτοια πρωτοβουλία πριν υπάρξει μια πραγματική στρατηγική για την καταπολέμηση της βίας. Και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στη συνάδελφο την κυρία Μπενίτα Φερέρο Βάλτνερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως γνωρίζετε, και βεβαίω δεν θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά, διότι ε, είμαι γυναίκα. Ε, είμαι, ε, με απασχολεί ιδιαίτερα η καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών και τη ε, απόκτηση δύναμη γενικότερα των γυναικών. Και αυτό όχι μόνο κατά τη διάρκεια τη θητεία μου ω επιτρόπου ε, αρμόδια για τα θέματα εξωτερική πολιτική, αλλά και στο παρελθόν, με, την, με την ιδιότητά μου τη Υπουργού. Να σα πω το εξή. Σε εξωτερικό επίπεδο, πέραν των ειδικών παρεμβάσεων στι χώρε στις ανεψόμενες χώρες, θέμα για το οποίο θα ε, μιλήσει ο φως μου ε, αργότερα, η εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών αυτή τη στιγμή αποτελεί σημαντικό άξονα της πολιτικής ε, υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική αυτή ενισχύεται και από τι συγκεκριμένε κατευθυντήριε γραμμέ που εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του 2008. Η υλοποίηση αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών διαρθρώνεται ε, σε, ε, σε τοπικό επίπεδο των τρίτων χωρών, εκεί όπου είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και μιλάμε για περίπου 90 τρίτες χώρες όπου οι, ε, ε, οι πρεσβείες μας αλλά και η αντιπροσωπεία της, Ευρω... αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναπτύξει το δικό τους πρόγραμμα δράσης για την υλοποίηση των κατευθυντηρίων γραμμών. Εκεί προβλέπεται μια ολόκληρη σειρά από πρωτοβουλίες για το χρονικό διάστημα 2009-2010 με συστηματικό τρόπο εμείς ε, θα εκπέμπουμε ένα σαφές μήνυμα. Η παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών δεν δικαιολογείται ε, με βάση τον ε, πολιτιστικό, την, την αρχή της πολιτιστικής σχετικότητας ή των παραδόσεων. Επίσης εμείς συνδέουμε την βοήθειά μας στις σχέσεις συνεργασίας και εκεί αναφερόμαστε συγκεκριμένα στα φαινόμενα εξάλληψης της βίας κατά των γυναικών και τη ενίσχυση των τοπικών θεσμών υπέρ τη ισότητα των δύο φύλων ή τη υποστήριξη ε, τη τροποποίηση τη νομοθεσία εκεί όπου προβλέπονται διακριτικέ μεταχειρήσει κατά των γυναικών. Γυναίκε, ειρήνη και ασφάλεια. Για για το 1325 και 18-20 ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών για την εφαρμογή αυτών των ψηφισμάτων. Και ε, το τρίπτυχο αυτό απαιτεί ολόκληρη μα την προσοχή. Ε, άλλωστε και εμεί ε, το Δεκέμβριο 2008 αποφασίσαμε μια συνολική προσέγγιση για την υλοποίηση όλων αυτών. Έτσι νομίζω ότι έχουμε ένα πυρήνα κοινών αρχών τόσο όσον αφορά τις επιχειρήσεις που άπτονται της ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, αλλά και όσον αφορά τις παρεμβάσει μας σε επίπεδο κοινοτικών μέσων. Αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει να μας επιτρέψουν να ενσωματώσουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο τη διάσταση γυναίκες στο σύνολο ε, των προσπαθειών αντιμετώπισης των συγκρούσεων από το, από το επίπεδο της πρόληψης μέχρι την επίλυση των ε, συγκρούσεων και την ανοικοδόμηση της ειρήνης σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο. Προσωπικά πιστεύω, ζήτησα την υποστήριξη 40 γυναικών που είναι ε, ηγέτιδες σε παγκόσμιο επίπεδο για την υλοποίηση του ψηφίσματος 1325 που όπως γνωρίζετε προτείνει τη διοργάνωση μιας υπουργικής ε, ε, διάσκεψης 10 χρόνια μετά από την, ιστορική, μετά από την ιστορική στιγμή της έγκρισής του. Και είμαι περήφανη γιατί συμφώνησε και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο κύριος Μπάνκιν Μουν, αλλά και κάτι άλλο και ίσως είναι πιο σημαντικό, θέλω να αναφέρω το γεγονός ότι προετοιμάζοντας αυτή την Υπουργική Σύνοδο όλο και ε, πιο μεγάλος αριθμός ε, διεθνών οργανώσεων όπως η Αφρικανική Ένωση αποφάσισαν να ενισχύσουν και να εντείνουν τις δικές τους προσπάθειες για την προώθηση ε, της εφαρμογής του ψηφίσματος 1325 κυρίως μέσω της ανάπτυξης εθνικών προγραμμάτων δράσης. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου με μια προσωπική νότα. Πρέπει να σας πω ότι εκτίμησα ιδιαίτερα αυτή την δυνατότητα οι πολιτικέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εσωτερικό και σε εξωτερικό επίπεδο να προσφέρονται ε, για την καταπολέμηση της βίας ε, εναντίον των γυναικών αλλά και για την υποστήριξη των γυναικών γενικότερα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι βλέπω ότι η δράση η οποία στο παρελθόν ήταν κάπω περιορισμένη και αφορούσε κάποιε προσωπικέ προσπάθειε, τώρα εντάσσεται απόλυτα μέσα σε μια απόλυτα κοινή προσπάθεια. Σα ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, ε, πρώτα από την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λογικού Κόμματος, η κυρία Ματέρα για 1,5 λεπτό. Sì, grazie Presidente. Σας ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Η εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο απαιτεί, απαιτεί σημαντική προσπάθεια και δέσμευση εκ μέρους όλων μας και των ευρωπαϊκών θεσμών και των κρατών μελών και της κοινωνίας των πολιτών. Η βία κατά των γυναικών πέραν του γεγονότος ότι αποτελεί κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οδηγεί σε βαρύτερες συνέπειες και σε τομικό και σε κοινωνικό επίπεδο που δεν μπορούμε να τις αγνοήσουμε. Γι' αυτό πρόκειται για ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε κάτω από διάφορες πτυχές σε πολιτιστικό επίπεδο. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την ιδέα ότι μπορεί δηλαδή να υπάρξει η παραμικρή δικαιολογία ε, της βίας αυτής με βάση ε, πολιτισμικές, κοινωνικές ή θρησκευτικέ ε, αρχές. Θα πρέπει να υπάρξουν εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ακόμα και στους νέους, δηλαδή στα παιδιά, μέσα στα ίδια τα σχολεία. Η διοργάνωση λοιπόν του Ευρωπαϊκού Έτους, όπως επαρελειμμένα έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα μπορούσε να έχει τη σωστή επίπτωση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο για να οικοδομήσουμε μια πιο συνεκτική και αποτελεσματική πολιτική. Σε πολιτικό επίπεδο θα πρέπει να θέσουμε το θέμα ανάμεσα στι προτεραιότητε τη πολιτική ατζέντα σε εθνικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θεωρώ λοιπόν σημαντικό και τελειώνω εδώ, να συνδέεται όλο και περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα Ηνωμένα Έθνη, έτσι ώστε να εργαζόμαστε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Και με αυτή την έννοια, ε, ε, ε, το γεγονός ότι υπήρξε η ακρόαση του Αντιπρόεδρου των Ηνωμένων Εθνών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν σημαντικό γεγονός. Θέλω λοιπόν να υπάρξει όλο και μεγαλύτερη συνεργασία εις όφελος όλων. Ευχαριστώ. Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Τόμσεν για μισό λεπτό. Tak, herr Kære kolleger, i dag Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα λοιπόν στις 25 ε, Νοεμβρίου έχουμε τη Διεθνή ημέρα των ε, Ηνωμένων Εθνών που αφορούν στην εξάλληψη της βίας εις βάρος των γυναικών. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο πρόβλημα στην κοινωνία μας που ε, δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί. Πρόκειται για το πρόβλημα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το δικαίωμα στην ασφάλεια και τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν ότι το πρόβλημα της ε, εσωτερικής βίας είναι ένα βαρύτατο πρόβλημα το οποίο στοιχίζει πολλές ε, περισσότερες ανθρώπινες ζωές από οποιοδήποτε άλλο ε, φαινόμενο όπως είναι ο πόλεμο, παραδείγματο χάρη. Είναι λοιπόν απολύτω απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει πάρα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καταθέσει ένα πρόγραμμα αγώνα ε, με οποιαδήποτε μορφή για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτών των γυναικών. Σε επίπεδο κρατών μελών είναι προφανέ ότι κανένα κράτο δεν θεωρεί ε, το πρόβλημα αυτό περισσότερο σημαντικό από κάποιο άλλο. Είναι αλήθεια ότι η Ισπανική Προεδρία ε, θεώρησε ότι η ε, μάχη αυτή κατά της βίας των γυναικών έχει πρώτη προτεραιότητα διότι συστήθηκε ένα παρατηρητήριο το οποίο εκλήθη να καταθέσει μια έκθεση που αφορά στη βία κατά των γυναικών και να διατυπώσει και προτάσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η βία. Η Ισπανική λοιπόν Προεδρία κατέθεσε μία πρωτοβουλία στο να συσταθεί ένα παρατηρητήριο το οποίο θα αποτελεί εγγύηση για, όλες, για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία ε, Παρβάνοβα για ένα λεπτό. Mr. President, dear colleagues, not only because... Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όχι μόνο λόγω του ότι σήμερα έχουμε αυτή τη Διεθνή Μέρα για την Εξάλληψη της Βίας, θα πρέπει γενικώ να θα κατά πόσο έχουμε κάνει αρκετά. Στην Ευρώπη η γυναίκα είναι αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης, ακροτριασμού των γενετικών οργάνων και βιασμών ε, σε περιόδου ε, πολέμου ο βιασμό χρησιμοποιείται και ω όπλο του εχθρού, όπω σημαίνει στο Κονγκό. Έχει λοιπόν φτάσει στιγμή να καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δράση που θα αντιμετωπίζει όλε τι μορφέ βία ει βάρο των γυναικών συμπεριλαμβανομένου και του σύγχρονου δολεμπορίου. Κυρία Επίτροπε, θέλω να σε ενημερώσω ότι σήμερα, κατά τη διάρκεια του ψηφίσματο για το πρόγραμμα τη Στοχόλμη, υπερψηφίσαμε μία τροπολογία που απαιτεί να υπάρξει πρόγραμμα δράση ε, για τη βία των γυναικών, να προστατεύονται τα θύματα ε, και να διώκονται οι δράστες. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτή τη φορά οι συναδελφοί μου και εσείς και το Συμβούλιο δεν θα παραθέσει και θα παραπέμψει στο θέμα της επικουρικότητας. Ελπίζουμε ταχύτατα να ε, δούμε να υπάρξει πρόγραμμα δράσης και ελπίζουμε το θέμα αυτό να παραπεμφθεί στην Ισπανική Προεδρία η οποία τάστε υπέρ αυτής της προτεραιότητας και ελπίζουμε αυτό να γίνει προτεραιότητα και για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος ομάδας των Πρασίνων, ο κύριος Ρωμέβα Ερουέδα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πράγματι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια σαφή νομική βάση για την καταπολέμηση όλων των μορφών βία κατά των γυναικών. Επίση, απευθύνω έκκληση προ το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ε, ε, ε, προχωρήσουν προ την κατεύθυνση τη χάραξη μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική προ την κατεύθυνση αυτή, ξεκινώντα από το ότι θα πρέπει να υπάρξει μηδενική ανοχή τέτοιων φαινομένων. Και αυτό πρέπει να έχει την προτεραιότητα για όλου του θεσμού. Το Κοινοβούλιο ζητά από, την, από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υπάρξει μια πιο συνεκτική πολιτική για την καταπολέμηση όλων των μορφών βία εναντίον των γυναικών. Και αυτό θα αποτελέσει ένα βήμα προ την ορθή κατεύθυνση. Επίσης, θα ήθελα να επενθυμίσω στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο το αίτημά μου για την αντιμετώπιση τη βία εναντίον των γυναικών ε, σε όλα τα θέματα σε παγκόσμιο επίπεδο ε, ε, όπου υπησέρχεται το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όσον αφορά τι σχέσει συνεργασία και αυτέ που ισχύουν και στι μελλοντικέ. Όπω αναφέρεται και στην έκθεσή μου. Ρωτώ λοιπόν την, Επιτροπή, την εκπρόσωπο τη Επιτροπή, μπορεί να πει δύο λόγια προ την κατεύθυνση αυτή. Επίσης, σας παραθέτω ε, στο παράδειγμα ε, του Κογκό ε, και σας λέω ότι αυτή τη στιγμή υπενθυμίζουμε το, ότι ο αγώνας είναι κοινό. χαιρετίζω λοιπόν και τους συναδέλφους που βρίσκονται στα πάνω, στις πάνω θέσεις, στους παρατηρητές που έρχονται από το Κογκό και σας λέω ότι ο αγώνας μας είναι κοινό. και η κυρία για λεπτά. Thank you. Violence against women, especially in the domestic environment. Η βία κατά των γυναικών, κυρίω στο περιβάλλον είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Και γι' αυτό ευχαριστούμε πολύ τον Πρόεδρο που το έφερε στο προσκήνιο. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτό δεν είναι ένα θέμα φίλων μόνο, δεν είναι θέμα ισότητο. Δεν είναι μόνο ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά είναι ένα θέμα ποινικού δικαίου καταρχήν και επειδή πρόκειται για θέμα ποινικού δικαίου, είναι θέμα κυρίαρχων κρατών και να πρόκειται στα κράτη-μέλη να αναλάβουν την πρωτοβουλία σύμφωνα με ε, τις στατιστικές πολλές γυναίκες θα ζήσουν αυτή τη βία στο σπίτι. Μπορεί να προλάβει αυτά ε, τα περιστατικά η Ευρωπαϊκή Ένωση με ευαισθητοποίηση και με την ευρύτερη συζήτηση για τη βία όχι μόνο κατά των γυναικών αλλά και των ανδρών. Σύμφωνα ε, με το Υπουργείο Εσωτερικών στη χώρα μας ένα σε έξι άτομα υποφέρει από γυναική βία. Πρόσφατα είχα συζητήσει ένα κέντρο προσφύγων γυναικών και, συζή... και ε, προέρχονταν από πολλές ε, κοινωνικές ομάδες. Δεν υπάρχουν στερεότυπα. Επηρεάζει η βία, το θύμα, την οικογένειά τους και τα παιδιά. Ε, καταστρέφει τις ζωές τους. Ο, ο, δρόμος για να αποκαταστεί τη ζωή τους είναι μακρύς και χρειάζεται υποστήριξη. Χρειάζεται ένας ε, ασφαλής χώρος να αποκτήσουν πάλι εμπιστοσύνη στον εαυτό τους για να λειτουργήσουν την κοινωνία. Αυτά τα προγράμματα χρειάζονται υποστήριξη και οικονομική υποστήριξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προλάβει με το να καταρρύψει ορισμένα ταμπού όσον αφορά ε, την βία κατά των γυναικών και των ανδρών. Είναι στο μέσο όπου εμεί ω κοινωνία δεν μπορούμε να γνωρούμε πλέον. Εξ των μη γεγραμμένων, η κυρία Στάσεν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, η κυρία Σβένσον έθεσε γραπτές ε, ερωτήσεις. Ε, η ε, Επιτροπή Γυναικών κατέθεσε επίσης ένα σχέδιο και εκεί αναφέρεται ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο επιτείνεται λόγω της ανισότητας μεταξύ των ανδρών και γυναικών. Το κόμμα για την ελευθερία δεν συμφωνεί απόλυτα με όλα αυτά. Βέβαια θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα, όμως όχι σε ευρωπαϊκό αλλά σε εθνικό επίπεδο. Γιατί το κόμμα για την ελευθερία ε, αποκηρύσει τη βία εις βάρος των γυναικών. Ε, σε μας ε, στην πατρίδα μας, διαπιστώνουμε φαινόμενα βίας εις βάρος μουσουλμάνων γυναικών διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν φαινόμενα όπως ακροτηριασμός των γεννητικών οργάνων των γυναικών. Ε, εμείς λοιπόν αποκηρύσουμε οποιαδήποτε μορφή βίας, κυρίως όμως αυτή τη βία που ασκείται εις βάρος των γυναικών μουσουλμάνων ε, θέλουμε να την προβάλλουμε γιατί είναι παντελώς απαράδεκτη. Ως εκ τούτου το δικό μου το κόμμα καλεί όλα τα κράτη-μέλη να ε, καταδικάσουν βαρύτατα και κατάφορα τη βία που ασκείται εις βάρος των μουσουλμάνων γυναικών. Köszönöm szépen, elnök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 Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω κάτι το οποίο ήδη ε, είπατε κι εσεί, ε, κύριε Υπουργέ. Σε μια πολιτισμένη κοινωνία δεν υπάρχει καμία θέση ή δικαιολογία για βία. Είναι η δέκατη η δεκατη επέτειο για μα, η δέκατη ευκαιρία για να θυμηθούμε τη δήλωση των ΗΠΑ για την ε, εξάλληψη τη βία εναντίον των γυναικών. η δέκατη λοιπόν επέτειο τη πρώτη διακήρυξη. Άκουσα του συναδέλφου, άκουσα και τα δικά σα και τι δικέ σα στην ομιλία και σκεφτόμουν τι θα συμβεί σε 10, σε 20 χρόνια. Αναρωτιόμουν για το κατά πόσο 10 χρόνια ή 20 χρόνια αργότερα ε, θα λέμε τα ίδια πράγματα ή μήπως η, ε, ε και, οι επόμενοι, αυτοί που θα μας διαδεχθούν θα υποστηρίζουν τα ίδια, ότι δηλαδή σε μια πολιτισμένη κοινωνία δεν, έχει, δεν υπάρχει θέση για βία. Ε, κοιτάξτε, ε, πρέπει να σας πω το εξή. Κοιτάξτε την κοινωνία μας. Θα δείτε ότι η επιθετικότητα όλο και αυξάνεται και δεν ισχύει το αντίθετο. Για κοιτάξτε την επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, γιατί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση εξάλληψη των φαινομένων αυτών. Και βεβαίως η οικονομική κρίση, διότι και αυτή έχει επιπτώσεις. Οι ψυχολόγοι θα το επιβεβαιώσουν. Η κρίση έχει αρνητική αρνητικέ επιπτώσει ανθρώπου και του αυξάνει την επιθετικότητα. Άρα το συνολικό θέμα τη βία εναντίον των γυναικών είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και ξέρω ότι πολλοί από του άρενε συναδέλφου μα υποστηρίζουν ότι και οι άνδρε είναι θύματα τη βία. Ναι, σωστό, αλλά δυστυχώ πρέπει να σημειώσουμε το, γυναικό, το, το γεγονό ότι οι στατιστικέ δείχνουν ότι το 55% των θυμάτων βία είναι γυναίκε. Δυστυχώ. Επίση, ε, ε, όσον αφορά το εμπόριο των ανθρώπων, και εδώ το 80% των, των ανθρώπων αυτών, των θυμάτων, είναι γυναίκε. Κύριε Πρόεδρε, ε, ε, κύριε Επίτροπε, ήρθε η στιγμή τα ευρωπαϊκά όργανα να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό με πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα. Περέζ, για μισή λεπτό. Κοιτάξτε, σήμερα εκατομμύρια ανθρώπων και γυναικών υψώνουν τη φωνή του ολόκληρο τον κόσμο για την εξάλληψη τη βία. Σήμερα δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μα να κλείσουμε τα μάτια απέναντι σε αυτό το πλήγμα τη σύγχρονη κοινωνία ε, που έχει να κάνει με σχέσει εξουσία ε, που έρχονται από το παρελθόν. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Δεν υπάρχει κανένα πρόσχημα. Γυναίκε δολοφονούνται σήμερα μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκε. Απέναντι σε αυτήν την πραγματικότητα όλοι είμαστε υπεύθυνοι. Τα ευρωπαϊκά όργανα, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, τα κράτη-μέλη και οι οργανώσει Όλοι θα πρέπει να ε, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα για να εξαλείψουμε το φαινόμενο αυτό. Για να προχωρήσουμε σε μια κοινωνία με περισσότερη ισότητα ε, και με αποφασιστική νομοθεσία προ την κατεύθυνση αυτή. Χώρε όπω η Ισπανία ανέλαβαν σαφή δέσμευση προ την κατεύθυνση αυτή. Ο νόμο ε, για, την, για την εξάλληψη τη βία λόγω φύλου αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Εκπαίδευση για την ισότητα των δύο φύλων, μέτρα πρόληψη, καταπολέμηση των στερεοτύπων, μέτρα νομικής αρρωγή και συνδρομής προ τα θύματα. Και θα μπορούσαμε να παριθμίσουμε παραδείγματα προ την κατεύθυνση αυτή. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό ε, η Προεδρία, η επόμενη, η Ισπανία, έθεσε ω βασική προτεραιότητα στην ατζέντα τη ε, την καταπολέμηση τη βία λογοφύλου και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει αποφασιστικά όλε τι πρωτοβουλίε που έχουν ως στόχο την κατεύθυνση αυτή. Ε, Α ενώσουμε τι προσπαθίε μα και την εργασία μα, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα βριστούμε στο πλευρό εκατομμυρίων γυναικών θυμάτων που δεν μπορούν να περιμένουν άλλο ούτε καν ένα λεπτό ακόμα. Κρέτου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Όπω υπόθηκε, η βία κατά των γυναικών είναι ένα πολύ σοβαρό φαινόμενο, το οποίο δεν έχει τύχει της αναγκαία προσοχής. Βεβαίως διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ορισμένες χώρες που πλήττονται περισσότερο επειδή βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Κάθε μορφή βίας, ιδίως σεξουαλική, εναντίον των γυναικών, των νέων γυναικών αλλά και των παιδιών, ε, έχουν φτάσει σε επίπεδα τρομακτικά σε χώρες όπως το Μπουρούντι, όπου υπάρχουν όμως και ορισμένες χώρες που χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλα ποσοστά βίας. Και η βία υπάρχει όμως και σε ήρεμες και δημοκρατικές χώρες. Γι' αυτό καθήκον μας είναι να καταστήλουμε αυτό το φαινόμενο και να κατεδικάσουμε ε, τους υπεύθυνους και να εξασφαλίσουμε την προστασία των γυναικών και να παράσχουμε όλη την απαιτούμενη υποστήριξη στα θύματα της σεξουαλικής βίας, ακόμα και γιατρική βοήθεια και τον τρόπο για την επανένταξή του στην κοινωνία. Τέλος, εν παρόδο θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή TV γιόρτασε ε, την ημέρα της, ε, Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο η οποία μας ε, παρουσίασε από το θέμα εδώ. Κύριε. Πρόεδρε, θα ήθελα να αφιερώσουμε αυτή τη Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη τη βία ε, στη μνήμη τη Άννα Πολιτόφσκα, για μια ε, δημοσιογράφου, μια γυναίκα που πλήρωσε με την ζωή τη, την αγάπη της για την αθλήτα, για την αλήθεια, συγγνώμη, στις γυναίκες της σε όλε τι γυναίκε που είναι θύματα τη βία. και ε, καταλαβαίνετε ότι αυτό ε, έρχεται ε, σε αντίθεση με τα στερεότυπα που προβάλλουν τα μέσα μαζική ενημέρωση για την εικόνα της γυναίκας. Όλα αυτά τα φαινόμενα οδηγούν σε καταπίνωση των γυναικών και αυτό είναι μορφή βία. Θα πρέπει λοιπόν να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να υπάρξει ένα συνεκτικό σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για στατιστικά στοιχεία, προσέχοντας ιδιαίτερα τους ανήλικους, τι ευάλωτε ομάδε, τι γυναίκε που είναι ευάλωτε όπω οι μετανάστριε κτλ. Θέλουμε όμω και συγκεκριμένα συγκεκριμένα παραδείγματα. Ε, αναφέρθηκε και η Επίτροπο με βάση τι κατευθυντήριε γραμμέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι γυναίκε στι ένοπλε συγκρούσει. Και να ε, ε, υποστηρίξουμε ακόμα και οικονομικά αυτά τα μικρά προγράμματα που προέρχονται από τι τοπικέ ε, οργανώσει και που προσπαθούν να ενσωματώσουν, να, ενσωματώσουν στην κοινωνία τι γυναίκε που είναι θύματα τη βία. Ξέρουμε ότι σήμερα έχουμε και νέε δυνατότητε με τη συνθήκη τη Λισαβόνα και με το πρόγραμμα τη Στοκχόλμη για να μπορέσουμε να καταστήσουμε αυτή την πολιτική πρόληψη εξή κοινοτική. Θα πρέπει όμω να αναφέρομαι και μια άλλη πτυχή. Ε, το γεγονό ότι η βία αυξάνεται σε επίπεδο ανηλίκων, σε επίπεδο νέων που συνδέεται με τα ναρκωτικά και με, το, και με την κατάχρηση αλκοόλ. Και θα πρέπει να μιλήσουμε για τα φαινόμενα αυτά, γιατί δεν μιλάμε αρκετά. Ευχαριστώ. Ε, σε για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εκατομμύρια γυναικών ε, υφίστανται βία, χτυπήματα, βιασμό και όλα αυτά απλά και μόνο γιατί είναι γυναίκες. Πεθαίνουν λοιπόν περισσότερες γυναίκες από τη βία που ασκείται εις βάρος τους από, τη, από γυναίκες που εθαίνουν από τον καρκίνο. Πρέπει λοιπόν να καταστήσουμε σαφές ότι στη σύγχρονη κοινωνία δεν υπάρχει χώρος ε, για τη βία. Αυτό πρέπει να το πούμε απέναντι στους πολιτικούς μας ε, ταγούς και πρέπει να το εκφράσουμε και απέναντι σε εκείνες τις ε, θρησκείες που εξακολουθούν να πιστεύουν ότι οι άνδρες είναι ανώτεροι. Στη δική μου τη χώρα η συντηρητική δεξιά περιέκοψε τα δικαιώματα γυναικών, είπε ότι οι γυναίκες να κάτσουν στην κουζίνα τους, ε, τελεία και παύλα. Ε, Κλησία, λοιπόν, κουζίνα <laughs> και γυναίκες. Οι γυναίκες εξάλλου ε, δεν έχουν και το δικαίωμα της τεχνητής γονιμοποίησης. Η γυναίκα λοιπόν καλείται να φέρει το σταυρό της στην Πολωνία και να δεχθεί και τον άνδρα που τη γρονθοκοπάει. Αυτό είναι μάστιγα στη σύγχρονη κοινωνία. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που ε, το Δεκέμβρη θα έχουμε εδώ μια συνδιάσκεψη στο Κοινοβουλίο μετά από πρωτοβουλία της Επιτροπής Γυναικών για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Uh, Δύο θέματα θέλω να σας πω αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτον, η μπλε κάρτα είναι για να υποβάλλετε ερωτήσεις ε, στον ομιλητή, όχι για παρεμβάσεις. Δεύτερον, έχουμε ήδη καθυστερήσει, είναι μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να δώσω το λόγο τουλάχιστον σε έξι άτομα, αλλά δεν μπορώ δυστυχώς σε παραπάνω. Θα δούμε βέβαια πώς θα πάει. Τώρα ε, στη διαδικασία του ΚΑΤΣΤΙΑΙ η κυρία Γκρούνη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κάθε μέρα στην Ευρώπη μια γυναίκα στι πέντε είναι θύμα βία. Η βία κατά των γυναικών είναι κάτι το απαράδεκτο, όποια και είναι η μορφή τη. Αλλά στην Ευρώπη ε, Πολλέ κοπέλε και γυναίκε ζουν μέσα σε ένα περιβάλλον εκμετάλλευσης ή επίθεσης. Είναι ανησυχτικά τα στοιχεία. Η επιθεση ειναι ανησυχητικα τα κατά των γυναικών έχει πολλέ μορφέ και εκδηλώνεται παντού. Ε, στο σπίτι, ε, κακοποίηση ακόμα και ε, μέσα σε, ε, στα ζευγάρια και είναι και τακτική πολέμου. Στην Ευρώπη η κονιακή βία είναι η πρώτη αιτία ε, θνησιμότητας για γυναίκες από 16 10-14 χρονών. Αυτή τη στιγμή συζητούμε αυτά τα θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και γυναίκες αυτή τη στιγμή είναι θύματα βιασμού. Θα πρέπει να αντιδράσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προστατεύει τον πιο ευαίσθητο πληθυσμό της η καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών είναι ο αγώνα κάτω των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα προγράμματα που υποστηρίζουν ε, τι ενέργειε ε, που έχουν αντικείμενο να αντιμετωπίσουν κάθε μορφή βία, δεν αρκούν. Πρέπει να ληφθούν νέα μέτρα για να υπάρξουν ευρωπαϊκά προγράμματα συνεκτικά. Υποστηρίζω την πρωτοβουλία ε, της οργάνωσης μιας ημέρα για την εξάρτηση τη βία αντί των γυναικών ε, που, που, υπάρχει στην, στην Ευρωκοινοβούλιο εδώ και 10 χρόνια. Είναι εδώ η κυρία Ροντζούλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ε, ε, θα ήθελα να αναφερθώ εγώ σε αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι Ματέρα και Στάσεν για, τις, ε, για το κατά πόσον η βία δικαιολογείται από πολιτιστικέ και θρησκευτικέ αρχέ. Θέλω να σα μιλήσω για μια προσωπική μου εμπειρία ω εθελόντρια σε μία από τι αποστολέ. Θα σα μιλήσω για την ιστορία μια γυναίκα τη Κάριν, μια γυναίκα που δεν ήθελε να φορέσει την μπουρκα. Ο σύζυγό τη για να την τιμωρήσει τη έριξε οξύ και το, το έκανε τη νύχτα, την ώρα που όταν ε, η γυναίκα αυτή. Τώρα η Κάριν φοράει την μπουρκα. Όχι γιατί θέλει να τη φοράει, γιατί αποτελεί επιλογή τη, αλλά για να κρύψει τα σημάδια αυτή τη ε, τρομερή βία που υπέστη. Λοιπόν, αυτή την ημέρα ελπίζω ε, να μην μείνουμε όλοι στα λόγια και απλά και μόνο να είναι άλλη μία ημέρα ε, που τη σημειώνουμε στο ημερολόγιο μα, αλλά να αλλάξουν πραγματικά τα πράγματα για τι γυναίκε αυτέ που είναι θύματα βία κάθε ημέρα. Τα λόγια λοιπόν να μετατραπούν σε πράξει και δράσει συγκεκριμένε. Ο κύριος Σταραμπέλα, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πολλέ είναι οι γυναίκε στην Ευρώπη και στον κόσμο που πολεμούν κάθε μέρα ε, για να εξαλειφθεί η βία εναντίον του. Αλλά δεν μπορούν μόνε του να διεξαγάγουν αυτόν τον αγώνα, διότι η βία κατά των γυναικών η οποία πραγματοποιείται σε συντριπτική πλειοψηφία από τους άντρε είναι και βία κατά της ανθρωπότητας και είναι φυσιολογικό και οι άντρε συμμετέχουν σε, αυτή, σε αυτόν τον αγώνα. Γι' αυτό ε, ε, θέλω να σας πω υπέρ τη καμπάνιας η οποία δημιουργήθηκε από άντρε και ξεκίνησε στον Καναδά πριν από 20 χρόνια κάποια μέρα ορισμένοι άντρε αποφάσισαν ότι είχαν καθήκον να παροτρύνουν άλλου άντρε να αντιμετωπίσουν τη βία κατά των γυναικών. Είναι η εκστρατεία Λευκή Κορδέλα. Επίση, ο αγώνα των γυναικών του Κονγκό κατά ε, της βίας εναντίον του που είναι καθημερινή και υπάρχουν ε, πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι πρέπει να μα συνδράμουν ε, κατά τη βία εναντίον των γυναικών υπάρχει σωματική αλλά και ψυχολογική βία και συχνά γνωρίζετε ότι τα λόγια πονάνε περισσότερο από του τακτικού χτυπήματα. Η κυρία Σάρμπου για ένα λεπτό. Um, Η βία εις βάρος των γυναικών στις ε, διάφορες μορφές της ε, είναι συνάρτηση του πολιτικοκοινωνικού πλαισίου. Μερικές φορές ε, πρόκειται για ψυχολογική κακοποίηση μέσα στην ίδια την οικογένεια, άλλες πάλι φορές χρησιμοποιούνται άλλες μορφές βίας. Όμως όλες αυτές οι μορφές ε, είναι απαράδεκτες κάτω από το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των δύο φύλων. Αυτές λοιπόν οι μορφές ε, βίας υπάρχουν σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Περισσότερα τα θύματα από αυτές τις μορφές βίας από ό,τι από τον καρκίνο. Και αυτό αγγίζει τον οτιό μυελό της κοινωνίας Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ενισχύσουμε τις ε, προσπάθειες μας αντιμετώπισης του φαινομένου. Και διαπιστώσαμε ότι η κακοποίηση όχι μόνο υφίσταται αλλά και αριθμητικά επεκτείνεται. Υπάρχουν πολλά ε, γεγονότα και στοιχεία που ε, αποκρύπτονται. Εγώ στη Ρουμανία τουλάχιστον αναφέρομαι και ισχύουν αυτά και στηρίζω την εκστρατεία των Εθνών για την αποκήρυξη της βίας εις βάρος των γυναικών. Η εκστρατεία αυτή έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία όσον αφορά τη βαρύτητα του προβλήματο. Σας Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η βία εις βάρος των γυναικών είναι έγκλημα ε, ανεξάρτητα με, το, με ποια μορφή πραγματοποιείται, είτε με εκβιασμό για γάμο, είτε με βιασμό, είτε με οτιδήποτε άλλο. Ειδικά αυτό που λέγεται για έγκλημα τιμή, είναι αυτό, απαράδεκτο. Εδώ δεν υπάρχει τιμή. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε για ε, να έχουμε το, ε, στο παράρτημα το Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Συνθήκη τη Λισαβόνα. Και εδώ, σε Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε ε, δεσμευμένοι να κάνουμε τα πάντα για να εξαλείψουμε τη βία. Επίση, αναφέρθηκε ότι η βία ε, στον πόλεμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ω όπλο του εχθρού, ο βιασμό πιο συγκεκριμένα. Και αυτό ε, συσχετίστηκε με το Κονγκό. Χρόνια τώρα συμβαίνει αυτό. Ε, βιασμό ε, μικρών γυναικών, μικρών κοριτσιών και γυναικών. Η κυρία Φέρερο Βάλτνε επισήμανε ότι όταν οι γυναίκες υπάρχουν στην κυβέρνηση, αυτό δεν σημαίνει ότι λύσαμε το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα δεν είναι των γυναικών, είναι όλων των ανθρώπων του κόσμου. Ως εκ τούτου, οφείλουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια στην Ευρωπαϊκή για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, όλο και περισσότερες ε, πρωτοβουλίε έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Δυστυχώς το φαινόμενο υπάρχει πάντα στην Ευρώπη και για κάθε ηλικιακή κατηγορία των γυναικών και για κάθε κοινωνική θέση της γυναίκας. Η βία κατά των γυναικών δεν είναι κάτι φυσιολογικό. Η βία κατά των γυναικών παντού στον κόσμο είναι έγκλημα παραβίαση του δικαιώματος ε, στην αξιοπρεπή ζωή, στην ασφάλεια ε, και στη σωματική και ψυχολογική ακαιρότητα. Εάν μιλάμε για βία, δεν πρέπει να παρουσιάσουμε τη γυναίκα μόνο ως θύμα. Αλλά η πράξη της βίας είναι ένα έγκλημα αυτό αυτό Δεν μπορεί να παραμείνει ατιμόρυτη. Και θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν όλοι για να γνωρίζουν τη δυσκολία αυτού του αγώνα. Senhor Presidente, que este Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres seja o início da queda. Στην προσπάθεια της εξάλληψης βίας εναντίον των γυναικών θα πρέπει να σταματήσει η σιωπή και διαφορία που υπάρχει στην κοινωνία μας. Αυτή είναι μια πραγματική πληγή ε, που ε, φύγει εκατομμύρια γυναικών. Η βία κατά των γυναικών είναι παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να συμμετέχει η γυναίκα στην πολιτική ζωή, στη δημόσια ζωή. Αλλά δεν μπορεί ε, με αυτόν τον τρόπο να είναι ε, η πολίτης ε, ίσης όρης με τους άλλους. Επίσης υπάρχουν διαφορετικές κουλτούρες και παραδόσεις που αυξάνουν τον ευάλωτο χαρακτήρα αυτών των γυναικών και τις περιθωριοποιούν, τις οδηγούν στη φτώγια, πράγμα το οποίο ε, τροφοδοτεί την εμπορία των γυναικών και την πορνεία πρέπει να υπάρχουν πολιτικά μέσα και ισχυρές πολιτικές για να μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία, να προωθηθεί η ισότητα των γυναικών και να υπάρξει ένα πραγματικό πρόγραμμα καταπολέμησης κάθε μορφής βίας εναντίον των γυναικών που θα συνοδεύεται από την εξάλληψη των διακρίσεων που υπάρχουν. Συγγνώμη από του εννέα ομιλητέ που παραμένουν. Τελευταία ομιλήτρια η κυρία Κιλ Νίλσεν για ένα λεπτό. Δεν είναι εδώ. Α, ναι. ε, Η δεκαετία του 2000 χαρακτηρίζεται από ε, επαγρύπνηση, περισσότερη, κρατήσεις, ε, ε πραγματικά ε, υπήρξε μεγάλη προσπάθεια, αλλά η βία κατά των γυναικών δεν μειώνεται. Το 2008, 156 γυναίκες πέθαναν ε, από το, λόγω, της, ε, λόγω της δράσης του συντρόφου τους. Ενώ είναι πάρα, μία στις δέκα είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Ε, πολλά μέτρα ε, λαμβάνονται, ε, οι κάμερες, τα βιομετρικά στοιχεία, αλλά όλα αυτά δεν μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της βίας που πλήττει τις γυναίκες σε όλες τις χώρες, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους τάξη, από την χώρα στην οποία ανήκουν. Αλλά στηρίζεται σε βία λόγω φύλου. Η σεξουαλική βία, όπως και ο ρατσισμός, συνίσταται στο να απαρνιέται κάποιο ε, το δικαίωμα ε, τη ύπαρξη του άλλου. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή απαιτείται μια ισχυρή και αποφασιστική πολιτική σε επίπεδο ενημέρωση, πρόληψη και προστασία. Να υπάρξει πολιτική βούληση για την εξάλληψη όλων των διακρίσεων, ε, στι οποίε, γιατί μέσα από τις διακρίσεις βρίσκει τις ρίζες στη η Πρέπει να υποστηρίξουμε ε, ε, ε, τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις γυναίκες και απαιτείται η κατάλληλη και η ακόλουθη πολιτική δέσμευση. Εξ ονόματος του Συμβουλίου για δύο λεπτά η κυρία Τόσενσον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. αξιότιμη κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής για την Ισότητα των Δύο Φύλων, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η βία λοιπόν μπορεί να ε, προσλάβει πολλές μορφές, όμως ο πόνος και τα βασανιστήρια ε, είναι τα ίδια για όλα τα θύματα. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι στον τομέα αυτό αναλαμβάνονται τόσες πολλές πρωτοβουλίες. Ελπίζω λοιπόν η ευρωπαϊκή συνεργασία να αποτελεί κινητήρια δύναμη για την αντιμετώπιση της βίας. Η συνεργασία μας πρέπει να είναι στρατηγικής μορφής απαιτούνται πρωτοβουλίες και δραστηριότητε και από εσά, διότι θέλω να επαναλάβω ότι η βία εις βάρος των γυναικών αποτελεί προτεραιότητα για τη Σουηδική Προεδρία. Πρώτον, στο πλαίσιο του προγράμματος της Οκχόλμης που θα εγκριθεί τους αμέσως επόμενους μήνες ε, γίνεται λόγος για το ότι ε, πρέπει να δραστηριοποιηθούν δραστηριοποιηθούμε περισσότερο για να αντιμετωπίσουμε τη βία εις βάρος των γυναικών. Κατόπιν, στις 2 Νοεμβρίου ε, η Προεδρία διοργάνωσε μια ημερίδα όπου η εκπρόσωποι μας ε, και τον ε, ε, κοινωνικών φορέων είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις για την αντιμετώπιση της βίας. Το φθινόπωρο εξάλλου είχαμε άλλο ένα συνέδριο που οργανώθηκε από την Προεδρία και εκεί επρόκειτο για τη βοήθεια προς όφελος ε, των ε, θυμάτων της βίας. Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε στις χώρες όπου υπάρχει σωματεμπόριο. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν ακόμα μπροστά μα πολλά εμπόδια αλλά οφείλουμε να μορφωθήσουμε όλοι να εξαλειφθεί η βία εις βάρος των γυναικών. Ε, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε ε, νίδη κατακλείδας να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση καθοριστικής σημασίας γιατί πρόκειται για βίες μορφές κατάχρησης και καταπάτησης ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όχι μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες, γιατί γίνεται πολλής λόγος ε, για το Κονγκό. Μάλλον θα πρέπει να μιλήσουμε και για άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, όπως ε, το Πακιστάν, παραδείγματος χάρη. Εχθές το βράδυ, μετά τη συνάντησή μας εδώ στο Κοινοβούλιο, είδα τις ειδήσει, είδα κάποιο πρόγραμμα στην τηλεόραση, στο κανάλι 24, και εκεί ε, γίνεται λόγος για την ε, κακοποίηση των γυναικών στο Πακιστάν. Απάνθρωπο, δεν μπορείτε να φανταστείτε, τραγικό. Όμως είναι και αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι, παραδείγματος χάρη, ε, Υπάρχουν τέτοια, αυτό που είπε μια κυρία συνάδελφος, ε, υπάρχουν περιπτώσεις όπως αυτή της γυναίκας που δεν ήθελε να φορέσει την μπουρκα. Σωστό αυτό. Είναι προφανές λοιπόν ότι η ε, σύγκρουση επιτείνεται, η κακοποίηση των γυναικών ε, χρησιμοποιείται ως ε, όπλο πολέμου και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα διαπιστώνει κανείς ότι ο κοινωνικός ιστός και η συνοχή παραδοσιακών κοινοτήτων καταστρέφονται και καταλήγουμε σε μια κατάσταση όπου έχουμε όχι μόνο επαναστατημένους αλλά και στρατιώτες και τους απλούς πολίτες οι οποίοι και αυτοί διαπράπτουν αυτά τα ιδεχθή εγκλήματα απάνθρωπα και εις βάρος των γυναικών και εις βάρος των παιδιών. Αρκετά μέλη ρώτησαν κατά πόσον θα ήταν δυνατόν να υπάρξει μια ευρωπαϊκή οδηγία. Ευρωπαϊκή λοιπόν οδηγία για τη βία εις βάρος των ε, γυναικών και για την δίωξη των δραστών. Δυστυχώς ε, θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει νομική βάση γι' αυτό. Υπάρχει κάποια νομική βάση στη συνθήκη της Λισαβόνας για συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να αναλυφθούν. Κυρίως όσον αφορά, όσον αφορά την εμπορία των γυναικών, την και εκμετάλλευση των παιδιών και την παιδοπορνογραφία. Εδώ πέρα υπάρχει σαφής αναφορά στις συνθήκες Λισαβόνα, αλλά η διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτή καθεαυτή δεν αποτελεί νομική βάση για να εκπονηθεί μια οδηγία. Νομίζω ωστόσο ότι η Επιτροπή πρέπει να εξακολουθεί, να εξετάζει, να διερευνεί πολλούς τομείς για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα, κυρίως με προγράμματα τα οποία όχι μόνο έχουν ως άξονα ε, την ανάπτυξη αλλά και ορισμένε ευάλωτε ομάδες αλλά επίσης και τα κράτη-μέλη. Επειδή και καθ' δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υποτίθεται αποτελεί παράδειγμα ε, στον κόσμο για τα, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των γυναικών, υπάρχουν πάντοτε προβλήματα. Μπορείτε να στηριχθείτε στην σημερινή Επιτροπή, αλλά και στην Προσεχή Επιτροπή, ότι θα συνεχίσει αυτές τις δράσεις, θα τις διευρύνει για τον απλούστατο λόγο ότι θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα αυτά τα μέτρα και όπως πρότεινε ένα μέλος, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν τις πρωτοβουλίες, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά, η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε κάθε επίπεδο και στα πλαίσια των ομοδιοτήτων μας πρέπει να έχουμε κατά νου αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ. Επίτροπε, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση πρέπει να σας πω ότι έχω λάβει διάφορε προτάσει ψηφίσματος εκ μέρου τη Επιτροπή Γυναικείων Θεμάτων ε, και ισότητα των Δύο Φύλων. Τώρα ολοκληρώθηκε η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Σα ευχαριστώ. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για μια πολιτική λύση όσον αφορά το φαινόμενο της πειρατείας στις ακτές της Ομαλίας.